Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την κοινή συζήτηση σχετικά με την κοινή εμπορική πολιτική. Το λόγο έχει κατά πρώτον για τέσσερα λεπτά η συγγήτρια, η κυρία Κουίστχαλτ Ρόβολ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πέτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζετε, ισχύς και δυνατότητα παρέμβασης και επιρροής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με την εμπορική πολιτική ε, αλλά και στη διαδικασία της υποδομής, δηλαδή κατά εξουσιοδότηση και, πράξεις και εκτελεστικές πράξεις, έχει ενισχυθεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας και ε, ως αποτέλεσμα αυτής της συνθήκης ε, πρέπει και στον τομέα της εμπορικής πολιτικής αλλά και στις αποφάσεις, δικασίες για λήψη σε δικασία αυτή, να ε, γίνει σχετική προσαρμογή στο νομοθετικό πλαίσιο. Το μεγάλο αυτό πακέτο λοιπόν μέτρων, το Omnibus 1, περιλαμβάνει πάνω από 20 κανονισμούς, μεταξύ των οποίων ο κανονισμός αντι-dumping και ο κανονισμός για την καταπολέμηση των επιδοτήσεων. Μετά από μακροχρόνια νομοθετική διαδικασία και πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου, μπορέσαμε τον Ιούνιο μόλις να καταλήξουμε σε μια πολιτική συμφωνία, συμβασμό. Δεν ήταν η διαδικασία απλή, αλλά μπορέσαμε εν τέλει να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα ήθελα να αναφέρω τώρα κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Και πρώτον, μέχρι πρόσφατα ο ρόλος των κρατών μελών την διαδικασία που αναπτύσσεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής για, το, για την καταπολέμηση του dumping και ε, των επιδοτήσεων ήταν αμφισβητούμενος και το, Συμβούλιο προσπαθούσε ακόμη περισσότερο με το μέτρο InfoPlus να το αμφισβητήσει. Το Κοινοβούλιο όμως με ε, επίκληση της συνθήκης Λισαβόνας ε, κατέθεσε προσφυγή, προσφυγή ε, διεκδικώντας ισότιμη μεταχείριση στην εμπορική πολιτική και απαιτούσε το Κοινοβούλιο τουλάχιστον τα κράτη-μέλη να μην ε, υπονομεύσουν με, με, με την ομοθεσία που θα εισηγούνταν το status quo. Έτσι λοιπόν, στην πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είδαμε ότι δεν ήταν καν ορατή η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε στην ε, τοποθέτησή μας αυτή όπου απαιτούμε να έχουμε τη δυνατότητα ε, να παραταθεί η διαδικασία αντι-dumping και κατά των επιδοτήσεων ε, στους 18 μήνες, τώρα είναι 15 μήνες η διάρκεια της διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό όμως ε, όταν ξεκινάει μια διαδικασία να ολοκληρώνεται βέβαια ως το δυνατόν πιο γρήγορα για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια για τους διαδίκους. Δεύτερο, τρίτον, με, όλες τις, με όλους τους κανονισμούς και τις ασφαλιστικές διαπιστώνουμε ότι ο πολιτικός ε, διακανονισμός με την ε, Κορέα ε, μετατρέπεται σε έναν κανονισμό που δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε. Η διαδικασία δηλαδή της επαλήθευσης μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στην τελική απόφαση όταν πρόκειται για προσωρινές ή ενδιάμεσες ρυθμίσεις μόνο η διαδικασία της διαβούλευσης εφαρμόζεται. Και έτσι αποφασίζει στη μία διαδικασία το Συμβούλιο και στην άλλη η Επιτροπή. Τα νομοθετικά κείμενα που, περιλαμβάνονται στο Omnibus και ο όγκος των μεταρρυθμίσεων που προτείνουν, των θεωρήσεων προτείνουν, οδηγεί στην απέτηση, στη διατύπωση της απέτηση για ένα πολύ πιο εύχριστο και ε, ολικό ε, μέτρο, για ένα γενικότερο δηλαδή νομοθέτημα, το οποίο θα εξασφάλιζε ε, ορατότητα στα κείμενα και περιμένουμε από την Επιτροπή μέχρι τον Ιούνιο του 2014 να, έχει καταθέσει αυτό το νέο κείμενο. Εν τω μεταξύ με το Omnibus και με τον εξυγχρονισμό της ε, προστασίας στις εμπορικές συναλλαγές, έκθεση ε, του κυρίου Γέλνερ δηλαδή, ε, είναι κάτι στο οποίο θέλω να αναφερθώ. Η ο κανονισμός Omnibus 1 αναφέρεται σε μια σειρά από κανόνες ε, κατά του dumping και των επιδοτήσεων, όπου προσαρμόστηκε μόνο η διαδικασία όμως και όχι η αρχή της προστασίας του εμπορίου αυτή καθεαυτή, ώστε να προχωρήσουμε κατά τρόπο λογικό ε, στον εξυγχρονισμό του μέσου για την προστασία του εμπορίου. Εν τέλει και συνολικά Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με, τους, ε, με το σεβασμό στον οποίο καταλήξαμε και ελπίζω ότι θα με υποστηρίξουν οι συναδελφοί στην Ολομέλεια. Μόνο μία πρόταση κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι ε, με συνέδραμαν στη συμπραγματεύση με το Συμβούλιο και την, με την Επιτροπή και κυρίως το Συμβούλιο, ιδιαίτερα το ΣΝΑΛΦΟ Λάιφριτ, γιατί έχουμε το Omnibus 1 και Omnibus 2 που προχώρησαν παράλληλα και μάλιστα μπόρεσαμε να τα διαπραγματευτούμε τα θέματα αυτά και να τα επεξεργαστούμε κατά τρόπο πολύ ε, συναδελφικό. Τον ευχαριστώ θερμά λοιπόν. Ευχαριστούμε κυρία Κουιστούτ. Για τέσσερα λεπτά τώρα έχει το λόγο άλλος εισηγητής, ο κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αλλά νομίζω το «gracias» θα είναι και τελευταία μου λέξη στα ισπανικά, διότι τα γερμανικά τα μιλάω καλύτερα. Δεν μπορώ παρά να ανταποδώσω τα συγχαρητήρια και την ευρωφροσύνη της κυρίας Ρόβολτ. Ήταν πραγματικά πολύ καλή η συνεργασία και την ευχαριστώ θερμά για τους λοιπούς συναδέλφους ε, που συνέβαλαν στα θέματα μας αυτά. Θέλω επίσης να εκφράσω θερμές ευχαριστίες και κυρίως θέλω να τιμήσω αυτούς των οποίων ποτέ δεν ακούγεται το όνομα, όλους αυτούς τους συνεργάτες της γραμματείας που έχουν κάνει και την πιο σοβαρή δουλειά, το πιο μεγάλο όγκο της δουλειάς. Ιδιαίτερα την κυρία Οκύφαλα και άλλους συναδέλφους που μας βοήθησαν πολύ. Η διαδικασία, η συνθήκη λοιπόν της Λισαβόνας έχει σαν αποτέλεσμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει αρμοδιότητες ε, συνομοθέτης στο εξωτερικό εμπόριο ε, και να συνδιαμορφώνει με τον τρόπο αυτό και τις ε, συμβάσεις διεθνούς εμπορίου. Έτσι λοιπόν και ενώ έχει υποτιμήθεί ο ρόλος συνθήκης της Λισαβόνας στο πεδίο αυτό, οδηγεί στο να έχουμε περισσότερη συμμετοχή στην εξωτερική πολιτική για το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος είναι κατά της συνθήκης Λισαβόνας, ταυτόχρονα πρέπει να ξέρει ότι είναι τα και κατά του εκδημοκρατισμού και τη ε, πρόσθεση περισσότερη διαφάνεια στην εξωτερική ευρωπαϊκή πολιτική. Πράγμα που βέβαια είναι λάθο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε να υλοποιηθεί αυτό το κομμάτι τη συνθήκη. Και για να επανέλθω στην ουσία τώρα, ο κανονισμό Omnibus 2 αναφέρεται στην επιτροπολογία, τη διαδικασία τη επιτροπολογία μετά την Λισαβόνα, την οποία μετατρέπει σε ένα σύγχρονο μέσο, με συναποφάση του Κοινοβουλίου. Έχει πέρασει αρκετό χρόνο, τέσσερα χρόνια ήδη που είναι υπερβολικά κατά την έποψή μου αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε ταχύτερα δυστυχώς. Ε, σημαντικό για μα τη διαδικασία αυτή, στην πραγματεύση αυτή και την αντιπαράθεση με το Συμφούλιο, σημαντικό ήταν ότι στις ε, κατεξοδότηση πράξεις μιλάμε για, λογική, για ορθολογικές προθεσμίες για την υποβολή των προτάσεων στο, Συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο και πρέπει ιδιαίτερα να επισημάνουμε, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, μπλέκεται στη διαδικασία ενός, ε, ενός κειμένου όχι μόνο με την αναπομπή του αλλά και κατά τη διαδικασία της εκτελεστικής πράξης κάτι το οποίο ξέρω ότι ίσως γέννησε κάποιες επιφυλάξεις για την Επιτροπή και το Συμβούλιο αλλά ήταν λάθος αυτό διότι αν γνωρίζει κανείς ποια είναι τα επιχειρήματα υπέρ και καλτά όταν έχει κανείς συμμετάσχει στην εμφάνιση των κατεξιοδότησης πράξεων τότε ασφαλώς βλέπετε ότι δεν είναι καθόλου περίπλοκη όλη αυτή η διαδικασία. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και έτσι σε συμφωνία με το Συμβούλιο ε, λέμε ότι θέματα κατεπήγοντα μπορεί να τα αναλαμβάνει σε αρμοδιότητες Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα υπόλοιπα όμως, για τα υπόλοιπα όμως πρέπει να στείλετε η γνώμη μας και νομίζω ότι εν τέλει το αποτέλεσμα στο οποίο καταλήγουμε είναι καλό. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι συνάδελφοι, ελπίζω και θα συμφωνήσω εδώ με τη συνάδελφο Κουίστου Θορόβολτ, ότι είναι μια καλή έκθεση, μια έκθεση η οποία θα εξασφαλίσει μια καλή και ευρία πλειοψηφία στην Ολομέλεια με την ψηφοφορία, θα βελτιώσει δε την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλέγμα. Υπάρχουν θέματα που μπορεί να μην σας φαίνονται πάρα πολύ ε, ενδιαφέροντα. Είναι όμως ε, θέματα τα οποία χρειάζονται πολλή δουλειά για να τα επεξεργαστούμε, τα οποία έχουν πολύ σοβαρές συνέπειες και τα οποία τελικά είναι πολύ σημαντικά. Και έτσι επηρεάζουν και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Νομοθέτη και μπορούμε νομίζω χάρη σε αυτά να καταλήξουμε σε ένα κανό, καλό ε, νομοθέτημα για την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Πολιτική Εμπορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Λάκφριτ. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα το λόγο έχει ο Επίτροπος Μιμικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο Επίτροπος Δεκούχτ δυστυχώς βρίσκεται σε υπουργική συνάντηση με τους ομολόγους μας από τον Ειρηνικό. Θέλω να ευχαριστήσω πάντως τους συζητητές, την κυρία Κίστουιτ Ρόβολ και τον κύριο Λάχτφριντ, όπως επίσης και τον καθηγητή Μορέιρα, πρόεδρο της Επιτροπής ε, ΙΝΤΑ, για την συνεργασία σας στον τομέα αυτό. Ενημερώνουμε τους κανόνες για τη λήψη αποφάσεων στην ε, εμπορική μας πολιτική υπό το φως κατεξουσιοδότηση πράξεων και εφαρμοστικών πράξεων έτσι όπως εισάγονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σημερινή συζήτηση προηγείται βέβαια της ψηφοφορίες για τη δεύτερη ανάγνωση. Είμαστε στο τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Μετά τον τελευταίο τριμερή διάλογο στις 5 Ιουνίου και την έγκριση στην Επιτροπή στις 11 Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα είναι έτοιμο να εγκρίνει την θέση του σε δεύτερη ανάγνωση. Το κείμενο που έχετε μπροστά σας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το αποτέλεσμα του τριμερούς διαλόγου που στηρίζεται απόλυτα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγκρίνοντας την θέση σε πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου, τελικά θα επιτρέψετε την θέση σε ισχύ την εφαρμογή του κειμένου. Φτάνοντα στο σημείο αυτό της νομοθετική διαδικασίας δεν ήταν εύκολο πράγμα. Μα πήρε χρόνο. Υπερβολικά πολύ θα έλεγα. Τρία χρόνια σχεδόν από την πρώτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την θέση σε ισχύ τελικά. Ε, Επίσης εκφράζουμε την λύπη μας επειδή χρειάστηκαν διάφορες παραχωρήσεις, αλλά χρειάστηκαν από όλε τις πλευρές προκειμένου να φτάσουμε σε συμβασμό. Σας ε, διαβεβαιώνουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδρασε όσο γίνεται πιο γρήγορα προκειμένου να καταλήξουμε στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε σήμερα. Θα ήταν επίσης σωστό να πούμε ότι με την έγκριση των δύο αυτών κανονισμών η Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική περνάει σε νέα αλλαγή. Με τη συνθήκη της Λεσεβόνας και τους κανόνες που διέπουν τις, εξου... τις εφαρμοστικές διατάξεις, καταλήγουμε σε μια νέα θεσμική ισορροπία που θα διέπει και τις κατεξοδότηση και τις εφαρμοστικές πράξεις στον τομέα της εμπορικής πολιτικής. Είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό. Με τις νέες αυτές διαδικασίες θα μπορέσουμε να δρούμε γρήγορα και να εφαρμόζουμε έτσι γρήγορα την ευρωπαϊκή εμπορική μας πολιτική. Θα είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Οι διαδικασίες λήψης απόφασης θα μας βοηθήσουν να κερδίζουμε χρόνο και άρα θα κερδίσουμε και αξιοπιστία στη διεθνή σκηνή. Θέλω επίσης να επιβεβαιώσω τις δηλώσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου. Ιδιαίτερα να σας πω ότι τώρα θα περάσουμε στην κωδικοποίηση των ε, λόγω κανονισμών με την ε, έκριση των δύο πακέτων. Όπως συμφωνήθηκε, η διαδικασία αυτή θα αρχίσει την 1η Ιουνίου του 2014 το αργότερο θα είναι πιο κατανοητό το πλαίσιο για όλους τους ενδιαφερόμενους. Τέλος, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά εκ μέρους του Επιτρόπου Τεγκούφτ, του συζητητές και το Κοινοβούλιο ολόκληρο για τη συνεργασία σας σε αυτήν την σημαντική υπόθεση. Θα προχωρήσουμε ώστε να λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο αυτό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Περνάμε τώρα στους ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Εκ μέρους του ΕΛΚ πρώτα απ' όλα για δύο λεπτά ο κύριος Κασπαρή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ θερμά την κυρία Κρίστου του Ρόβολτ και τον κύριο Λάιχφριτ. Ήταν πολύ καλή δουλειά που έκαναν τους τελευταίους μήνες σε συνεργασία με τους κοιόδους εισηγητές και χαίρομαι ιδιαίτερω που μπορούμε φέτος ακόμη να κλείσουμε το θέμα αυτό. Για τις ε, κατεξοδότητες συμπράξεις λοιπόν ε, δίνουμε την δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλαμβάνει νομοθετική πρωτοβουλία και αυτόνομα μόνη τη, δηλαδή σε ορισμένε περιπτώσει και υπό ορισμένε συνθήκε. Αυτό όμω σημαίνει και περισσότερε ευθύνε για όλου μα. Πρέπει και εμεί ω νομοθέτη, γιατί σε κάθε ε, θέμα, όπω και στον τομέα του εμπορίου, πρέπει να αναλογιζόμαστε τι επιδιώκουμε, ποιε είναι οι λεπτομέρειε για τι οποίε μπορούμε να αφήσουμε ένα περιθώριο χειρισμών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό νομίζω θα πρέπει να μα απασχολεί σε επόμενε εβδομάδε πολύ εντατικά. Για την Επιτροπή ταυτόχρονα σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλογίζεται τι θα ρυθμίσει με τι κατεξουδότηξει πράξει και πόσο λεπτομερώς και νομίζω ότι σε αντίθεση με άλλα εγχειρήματα για το αν ε, θα απαγορεύεται το ένα ή το άλλο συστατικό ή το ένα ή το άλλο είδο σκεύου. Ε, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί η Ευρωπαϊκή σκευου νομιζω οτι στην περιπροκειμενη περιπτωση μπορει η ευρωπαικη επιτροπη να ε, δώσει απαντήσεις. Και επίσης πρέπει ως ελεκτικό όργανο να αναλογιστούμε και πάλι για το μέλλον τι είδου ε, κατεξουδότηση πράξης θα αποδεχόμαστε για, την, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποια ζητήματα θα ζητούμε να διευκρινιστούν σε άλλο επίπεδο και σε ποια θα θέλουμε να συστήσουμε διεξοδικά και εν ώψη της αυριανής όπου θα κληθούμε να ψηφίσουμε για κατεξουδότηση πράξης. Προφανώς, εάν δούμε ας πούμε το σύστημα γενικεφανοπροτηρημίσεων προτιμήσεων ε, plus ε, και τις κατεξουδότητες συμπράξεις νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια καθαρή ιδέα του τι θα αφορούν αυτές οι στην συμπράξεις. Πάντως νομίζω ότι είναι πολύ καλό γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε επιπλέον αρμοδιότητες σε ένα πολύ σημαντικό τομέα που είναι το εξωτερικό εμπόριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κασπαρή. Εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα για δύο λεπτά ο κύριος Μορέιρα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Κάσπαρη είπε επιτέλους. Μετά από τέσσερα χρόνια, αφού το άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας, το νομοθετικό πακέτο ομνημούς 1 και 2 επιτέλους ευθυγραμμίζονται με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε θέματα καταξουσιοδότηση πράξεων και εφαρμοστικών πράξεων. Είναι μια μικρή επανάσταση της συνθήκης της Λισαβόνας αυτό. Χρειάστηκαν όμως τέσσερα χρόνια για να ευθυγραμμιστούμε με τη συνθήκη. Είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πήρε υπερβολικά πολύ χρόνο. Η καθυστέρηση αυτή στη νομοθετική διαδικασία είναι ένα μάθημα που πρέπει να πάρουμε για να αποφύγουμε την επανάληψη στο μέλλον το Συμβούλιο θα πρέπει να τροποποιήσει και εκείνο τις διαδικασίες για να μπορέσει σε εύλογο χρονικό διάστημα να μπορεί να δίνει απαντήσεις στους Ευρωπαίους πολίτες. Από την πρώτη στιγμή η εντολή διαπραγματεύσεων πρέπει να είναι ευέλικτη. Και ακόμα και αν ψηφίζουμε εδώ στην Ολομέλεια χρειάζεται ευελιξία στις διαπραγματεύσεις. Είναι αναγκαίο στις διοργανικές διαπραγματεύσεις. Πρέπει να αποφύγουμε τις άκαμπτες διαδικασίες. Καταφέραμε πάντως να φτάσουμε σε μια ικανοποιητική συμφωνία. Διατήρησε τις αρχές του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διάφορα ζητήματα, όπως για την διάκριση ανάμεσα στις κατεξουσιοδότηση πράξη και εφαρμοστικές πράξεις. Είναι πολύ σημαντικό που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τον έλεγχο της πρώτης κατηγορίας. Πολύ σημαντικό επίσης και για την συμβουλευτική διαδικασία και την εξέταση σε επιτροπολογία. Επίσης, επεκτάθηκε και προθεσμία για να μπορεί να υποβάλει ένσταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφόσον υπάρχουν και πολιτικά στοιχεία. Ήταν μια περίπλοκη νομοθετική διαδικασία. Και εδώ δημόσια, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές μας. Τους ευχαριστώ για την ε, δέσμευση που ανέλαβαν και θέλω να ευχαριστήσω και την ε, Προεδρία του Συμβουλίου που μας βοήθησε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για το πνεύμα συνεργασίας σας προκειμένου να καταλήξουμε σε λύσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μορέιρα. Εκ μέρους των φιλελεύθερων για δύο λεπτά τώρα έχει το λόγο ο κύριος Ρινάλντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο καθηγητής Μορέιρα, πρόεδρος της Επιτροπής μας, έχει δίκιο. Τέσσερα χρόνια για να καταλήξουμε σε αυτό το σημείο είναι μάλλον υπερβολικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους εισηγητές που επιτέλους κατάφεραν να περατώσουν αυτό το τριμερή διάλογο και αυτή τη συμφωνία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Σε τελική ανάλυση με βάση τις νέες αρμοδιότητες ε, θα μπορούσαμε να φτάσουμε πιο νωρί ε, σε ό,τι αφορά τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Πέρα όμως από όσα συμφωνήθηκαν και που βρίσκουν σύμφωνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτη συνείδηση ότι θα πρέπει να γίνουν πολλά, όχι μόνο μέσα από τους κανόνες, αλλά και μέσω του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας εμπιστοσύνη που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου και αυτό σε ό,τι αφορά το Κοινοβούλιο, αλλά και από την αντίθετη πλευρά. Πιστεύω ότι πάντοτε καταφέραμε να συνεργαστούμε <coughs> με απόλυτη συνέστηση της ευθύνη μας και σε ό,τι αφορά ορισμένα πρόσφατα συμβάντα, σκέφτομαι το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων Όσο προς 9-10 ε, δικαιούχους ε, χώρες, ενδεχομένω η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη αίσθηση συνεργασία. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αυτή διαβούλευσης όπως έχει συμφωνηθεί είναι αναγκαία και είναι αναγκαία για δύο λόγους. Από τη μία πλευρά, δίχως άλλο, το γεγονός ότι κινούμεθα με ταχύτερους ρυθμούς και δεύτερον δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από τις διαθεσμικές σχέσεις υπάρχουν ολόκληρες επαγγελματικέ κατηγορίες, υπάρχουν οι λεγόμενοι stakeholders οι οποίοι αναμένουν τα αποτελέσματα των εργασιών μας και οι οποίοι θα πρέπει να πούν την άποψή τους και που χρειάζονται μια διαδικασία η οποία να τους εμπλέξει όσο γίνεται περισσότερο. Από αυτή την άποψη το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρινάλντι. Περνάμε στους υπόλοιπους ομιλητές. Για δύο λεπτά ο κύριος Ιακολίνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τέλος καλό όλα καλά, όπως είπαν οι συναδελφοί μου στις παρεμβάσεις του. Χάρη ε, στην ε, αφοσίωση των δύο ε, εισηγητών. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι φτάνουμε, είμαστε τώρα στην τελευταία φάση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει μια πραγματική δέσμευση σε ό,τι αφορά τον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων θα απαιτήσει νέε και σαφώ καθορισμένες ευθύνε. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών μας. Υπάρχει ανάγκη να ενδυναμώσουμε την εμπορική μας πολιτική και αυτό θα πρέπει να γίνει σε στενή συνεργασία με άλλους σημαντικούς φορείς. Το TDI για παράδειγμα ε, με το οποίο Ελπίζουμε να, έχουμε μια, να δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία ανάπτυξης στις ευρωπαϊκές εταιρείες για να μπορέσουν να αντισταθμίσουν τη ζημία που έχουν υποστεί, απλοποίηση, διαφάνεια των διαδικασιών και για τους εισαγωγείς και για τους εξαγωγείς για να υπάρξει πλούτος γιατί αυτό θέλει στη συνθήκη της Λισαβόνας εστιάζοντας κυρίως στην εμπορική πολιτική. Ο βασικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρξει ένα νομοθετικό πλαίσιο είναι σημαντικό. Για να υπάρξουν ενιαίοι κανόνες και αυτό είναι κάτι που μας βρίσκει σύμφωνος. Μια εμπορική πολιτική η οποία οποία θα εγγυηθεί την ανταγωνιστικό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, δεχόμαστε λοιπόν με χαρά τις δύο συστάσεις γιατί υπαγορεύουν σαφείς κανόνες σε ό,τι αφορά αντισταθμιστικές εισφορές και κωδικοποίησεις και συνεπώς βοηθούν την εμπορική πολιτική. Αυτό ε, μας χρειάζεται να εξαλείψουμε τις αθέμητες πρακτικές και να εγγυηθούμε στις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα διεθνές ανταγωνιστικό πλαίσιο σύμφωνα ενιαίους κανόνες. Ένα κοινοβούλιο όλο, που θα έχει όλο και πιο κεντρικό χαρακτήρα και θα μπορεί να εγγυηθεί διεθνείς συμφωνίες και ένα πλαίσιο πολύ πιο, πιο απλοποιημένο και θα δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες για ένα διεθνές εμπόριο που οι ε, ε, κανονισμοί ε, επικεντρώνουν τον κεντρικό χαρακτήρα του κοινοβουλίου μα. Ευχαριστούμε κύριε Κολίνο. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Catch ένας μόνο έχει ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Μπάνκι. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι. Στα ουγγρικά λέμε το καλό αργεί να γίνει. Βλέπουμε όμως ότι μπορέσαμε επιτέλους να ολοκληρώσουμε αυτά τα καλά νομοθετήματα. Τέσσερα χρόνια χρειάστηκαν. Πολύς χρόνος. Αλλά ήταν αναγκαίο να προχωρήσουμε με σύνεση και προσοχή. Και ελπίζουμε ότι με τους νέους αυτούς βασικούς κανόνες θα μπορέσουμε να δείξουμε και ευελιξία περισσότερη και αποτελεσματικότητα. Αυτό το χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Ιδάλλως άλλω ε, θα βρισκόμαστε σε μειονεκτική σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας αυτό το μεγάλο αγώνα του ανταγωνισμού. Νέε ρητρε λοιπόν και μέτρα προστασία, Αναμένουμε να δούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλού τομεί έχει νέε και ευρείε αρμοδιότητε, και είμαστε βέβαιοι, ελπίζουμε μη τι άλλο, ότι θα μπορούμε και να ε, ελέγχουμε τι δραστηριότητε της Ευχαριστούμε. Επίτροπο τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ κύριε Μιμικά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Δεν θέλω βέβαια να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι εγκρίνοντα αυτή τη διοργανική συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορεί πλέον να αντιδράει πιο καλά για να υποστηρίζει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, διότι μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερο την πιο στενή συνεργασία με τα άλλα όργανα. Υιοθετώντα τι ρυθμίσει αυτέ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπει στην εφαρμογή των νέων κανόνων ήδη από την αρχή του 2014 και στην ενεργοποίηση των νέων διαδικασιών και καναλιών μέσα στα πλαίσια τη νέα αυτή συμφωνία με νέε δομέ. Θα μπορέσουμε να ελέγχουμε την λειτουργία του συστήματος προκειμένου αυτό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και περισσότερο κατανοητά για τους πολίτες μας. Τέλος. Θέλω να υπογραμμίσω την εκτίμησή μας στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο αντιλήφθηκε το κατεπήγον των δύο αυτών θεμάτων τώρα μάλιστα που είμαστε σε έντονη νομοθετική δραστηριότητα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Κουίστοτ Ρόβολ. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, για την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό βεβαίω να είναι δημοκρατικές οι για στι αρμοδιότητες για το εξωτερικό εμπόριο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη την Ήπειρο. Δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω περισσότερο τη σημασία. Και θα ήθελα με μια πικρή ηρωνία να πω ότι κράτησε πάρα πολύ όλη αυτή η διαδικασία μέχρι ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιδράσει γιατί θέλει να, αλλάξει, να τα κρατήσει όλα όσο όπως είχαν ενώ το Συμβούλιο διεκδικούσε επιστολές αρμοδιότητες και όλοι οι υπόλοιποι διερωτούνταν γιατί τώρα το Κοινοβούλιο θέλει να ε, διεκδικήσει τις ε, αρμοδιότητες που προβλέπει η συνθήκη γιατί αυτό λέγαμε Και εν τέλει φτάσαμε σε αυτή τη συμβαστική λύση. Καλό. Και σημαίνει ταυτόχρονα ότι έχουμε δουλέψει καλά μαζί. Κύριε Επίτροπε, και απευθύνω θερμές ευχές στον κύριο Ντεγκούχτ, είπατε ότι η Επιτροπή θα μπορεί να, διαδραματι... να δράσει πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Ναι, αυτό ήταν πάντα και το μέλημά μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για το Omnibus. Μπορεί και οφείλει. Αλλά το Κοινοβούλιο θα παρακολουθεί καλύτερα και θα ελέγχει καλύτερα την εκτέλεση από το εκτελεστικό όργανο και βεβαίως με κάθε φιλική διάθεση αυτό το κοπιαστικό καθήκον θα το αναλάβουμε και θα το εκτελέσουμε. Ευχαριστώ την κυρία Κουίστχολτ. Κλείνει αυτό το γύρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, η πολιτική εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχει ανοίξει νέους ορίζοντες και πανιά. Είναι πιο δημοκρατική, πιο κοινοβουλευτική. Η Επιτροπή τώρα ε, θα ελέγχεται πολύ πιο προσεκτικά ε, μας λέτε κύριε Επίτροπε ότι θα, δρά, θα δράτε πιο γρήγορα. Ναι, αλλά και εμείς πολύ πιο γρήγορα θα πατάμε το φρένο όταν δεν αντιστοιχούν όσα, όσα πρέπει αυτό που κάνετε. Και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι η εμπορική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι και κοινωνική πολιτική και πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και περιβαλλοντική πολιτική. Γιατί το καταφέραμε να είμαστε εμείς αρμόδιοι, να μεριμνούμε εμείς η ευρωπαϊκή πολιτική εμπορίου να διαμορφωθεί κατά τρόπο διαφορετικό από ό,τι μέχρι τώρα. Και πολύ καλό το βρίσκω αυτό. Αυτό είναι και ο σωστός δρόμος πιστεύω σε, μια, σε ένα μέλλον διαφορετικό πια για την εμπορική μας πολιτική. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ψηφίσουμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Επόμενο σημείο.